Herr Präsident! Die am 2. Februar 2012 unterbrochene Sitzung. Ξεκινάει και γίνεται επανάληψη της Συνόδου. Σας παρακαλώ να καθίσετε. Το πρωτόκολλο Τη συνεδρίασης τη 1ης και 2ης Φεβρουαρίου και τα εγκεκριμένα κείμενα τα έχετε λάβει. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις θεωρούμε ότι τα πρακτικά λοιπόν εγκρίνονται ούτως. zuständigen Behörden des Vereinigten Königreiches haben mir mitgeteilt, dass Frau Οι αρμόδιε αρχέ ε, του Ηνωμένου Βασιλείου μου ανακοίνωσαν ότι η κυρία Ελίζα Βεθλίντ θα αντικατασταθεί από τώρα, τον, από 6 Φεβρουαρίου του 2012, από τον κύριο Φίλιπ Μπενιόν. Τον καλωσορίζω. Είναι εδώ ο κύριος Μπενιόν. Πού είναι? Herr Benjen, herzlich willkommen. Σας καλωσορίζουμε στο Κοινοβούλιο. Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Geschäftsordnung ich erinnere daran dass jedes mitglied mit vollen rechten an den sitzungen des parlaments und seiner organe teilnimmt solange sein mandat nicht geprüft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 τον κύριο Γύρι Μασάλκα και τον κύριο Ρίκο Περόνι τους όρισα ως ε, αναπληρωτές ε, από τους ομάδες του ΕΛΚ, του ΑΛΔΕ, των Πρασίνων και της ΓΚΟΥΝΕ και των μη εγγυγραμμένων. Έλαβα ε, υποψηφίους και ο κατάλογος θα δημοσιευτεί στα πρακτικά. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίνονται αυτές, αυτοί οι διορισμοί να σας ανακοινήσω ένα, μια ανακοίνωση βάσει του άρθρου 2016 να σας διαβάσω δεν σας διαβάσω τους τίτλους αλλά σας παρακαλώ να κοιτάξετε στο ίντερνετ ε, το Seance Direct και να διαβάσετε τα σχετικά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 Στην Δευτέρα δεν έχουμε αλλαγές για την ημερήσια διάταξη. Θα παραμείνει όσο έχει η πράσινη τώρα. Ζήτησε για να γίνει συζήτηση για, τα, για τις αμόλογα σταθερότητα μετά τη συζήτηση ε, για το Μαρόκο. Ζητάει κανείς από, το λόγο, από τις πρασίνες το λόγο. Όχι. Σωστά το είπατε. Θέλουμε επειδή είναι τρεις εκθέσεις και συζήτησεις από την Επιτροπή Αγροτικών Ζητημάτων να συζητηθούν μαζί. Θέλουν λοιπόν οι πράσινοι να συζητηθεί το θέμα για τα ομόλογα σταθερότητα μετά τη συζήτηση για ε, το Μαρόκο, για την Ευρωπαϊκή Συμφωνία.